Συνάδελφοι, ήδη έχουμε καθυστερήσει. Οπότε ας πάμε στο σημείο 2 που είναι το σχέδιο της διάταξης για σήμερα. Νομίζω πως μπορούμε να το εγκρίνουμε και επίσης μπορούμε να δούμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου. Τώρα έχω κάποιες ανακοινώσεις να σας πω ότι Η γραμματεία μας είναι εκπληκτική, έχει ήδη τελειώσει τη συνόψηση του 2000, των αναφορών του 2015 και θα λάβετε τα τελευταία έγγραφα αυτή τη βδομάδα για να τα εξετάσετε και για να αποφασίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι η καθυστέρηση που είχαμε μαζευτεί μικραίνει όλο ένα μέρα με την ημέρα και μέχρι το τέλος του έτους δεν θα έχουμε πια καμία καθυστέρηση. Τα ακούσατε αυτό κύριε Βαλέσα. Με προσέξατε τι σας είπα κύριε Βαλέσα. Κύριε Βαλέσα είπα ότι η καθυστέρηση υποθέσεων που είχαμε μειώνεται και μειώνεται και προς τα τέλη του έτους θα έχουμε καλύψει τελείως την καθυστέρηση. Η γραμματεία μας λοιπόν κάνει εξαιρετική δουλειά. Τώρα, για τα θέματα που είναι στο, στη λίστα Β και για το διαδικασία που συμπεριλαμβάνεται στις κατευθύνσεις γραμμές θα σας θυμίζω ότι το κλείσιμο ε, αναφορών στη κλίστα Β βασίζεται σε ήδη υπάρχουσες ανακοινώσεις από την Επιτροπή μας ή άλλα ή από την Επιτροπή ή άλλα έγγραφα. Όταν λοιπόν ζητάτε για περαιτέρω ενέργειες, ελέγξτε πρώτα στο ΙΠΕΤΗ, αν οι ενέργειες που ήδη έχουν γίνει αρκούν ή όχι για τη συγκεκριμένη αναφορά. Γιατί κάποιες φορές ζητάμε περισσότερες πληροφορίες, ενώ όλες οι πληροφορίες ήδη υπάρχουν. Αλλά δεν τις έχουμε ελέγξει προκαταβολικά. Έχουμε το σημείο διάφορα, δεν έχει ζητήσει το λόγο εκεί κανείς και στο σημείο 6 με χαρά θα εξετάσουμε την αναφορά την αριθμό 1270 1270-2014 σχετικά με τη χειραγώγηση όσον αφορά τηλεοπτικές άδειες. Ο κύριος Γιάννη Λουθεράν που είναι ο αναφέρον είναι μαζί μας και σας δίνω το λόγο για 5 λεπτά κύριε Λουθεράν. Καλωσορίσατε. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Okay. Thank you. Ε, εντάξει, σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα σλοβακικά, δεν υπάρχει πρόβλημα, ελπίζω. Ωραία. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι Ευρωβουλευτές, καταρχάς ε, στείλαμε αυτή την αναφορά ε, γιατί δεν ήξερα αν ε, γνωρίζετε την υπόθεση αυτή. Είδαμε το αρχικό κείμενο της αναφοράς βρίσκεται στη Σλοβακία στο και γιατί είναι συνταγματικό δικαίωμα των Σλοβάκων πολιτών ε, να εκπέμπουν ελεύθερα ε, σε τηλεοπτικά κύματα ε, και έχει παραβιαστεί. Το 2012 δια νόμου οι πολίτες υποχρεούνται να πληρώνουν για τη δημόσια τηλεόραση, πράγμα που παραβιάζει το δικαίωμα των πολιτών. Η σύνδεση στη τηλεόραση καταγράφεται, ωστόσο, η εταιρείε δεν μπορούν να καλύψουν όλη την επικράτεια της Σλοβακίας με ε, εκπομπές δημόσιας τηλεόρασης. Ε, σε πολλές περιοχές οι πολίτες καθιστούν ε, απλούς μηχανισμούς για να μπορούν να, να, να λαμβάνουν το σήμα. Σε άλλες περιοχές όμως είναι υποχρεωμένοι να έχουν δορυφορική σύνδεση, η οποία δορυφορική σύνδεση παρέχεται από κρατική εταιρεία δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στις εκπομπές, όμως εκεί δεν υπάρχει κανένα έλεγχος και καμία εποπτεία. Δόθηκε μάλιστα σε ιδιωτική εταιρεία και η εταιρεία αυτή τρομοκρατεί τους πολίτες, οι οποίοι εάν δεν πληρώσουν τη χρέωση τότε μπλοκάρτε το σήμα από την ιδιωτική αυτή εταιρεία, η οποία μάλιστα εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Χρησιμοποιεί και χειραγωγεί στοιχεία η ίδια εταιρεία και χρησιμοποιεί και άλλες εταιρείες στην Σλοβακία και στην Τσεχία, ώστε να αναγκάσει τους πολίτες να πληρώνουν για ε, τις εκπομπές. Ε, η αρχή λοιπόν της ουδετερότητας παραβιάζεται, καθώς και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η εταιρεία αυτή στέλνει επιστολές οι οποίες ε, δεν στέλνονται καν με συστημένες επιστολές. Και πολλές φορές έχει γίνει χειραγώγηση των στοιχείων των πολιτών. Δηλαδή, οι πολίτες αναγκάζονται να πληρώνουν τόσο για τη δημόσια τηλεόραση της Σλοβακίας, όσο και για την ιδιωτική αυτή εταιρεία, η οποία δηλώνει ότι έχει έδρα στο Λουξεμβούργο και άρα μόνο λουξεμβουργικές αρχές μπορούν να την ελέγξουν. Εν τω μεταξύ, κάποιες φορές αυτή η ίδια εταιρεία αλλάζει τις παραμέτρους στις κάρτες Τη δορυφορική τηλεόραση και αν ο πολιτή δεν παρακολουθήσει τηλεόραση, α πούμε γυρνώντας από διακοπές, ε, το σύστημα είναι μπλοκαρισμένο και αν θέλει να διαμαρτυρηθεί ο ίδιο ε, για το μπλοκάρισμα αυτό πρέπει να καλέσει έναν ε, τηλεφωνικό αριθμό επιπληρωμή και μάλιστα από πολύ μεγάλη πληρωμή και είναι και πολύ δύσκολο να έχει πρόσβαση σε άνθρωπο, σε συνομιλητή ακυρώνονται δε οι κάρτες και οι πολίτες πρέπει να ε, αγοράσουν νέες συνδρομητικές κάρτες. Πρέπει να δεχτούν δε πολύ κακούς όρους και προϋποθέσεις. Το κράτος δεν πληρεί την αποστολή του και τη λειτουργία του, γιατί οι Σλοβακικές Εθνικές Αρχές έχουν ενημερωθεί για αυτό το θέμα, τους έχει κοινοποιηθεί, ωστόσο δεν έχουν κάνει τίποτα. Πρόκειται για ένα καρτέλ το οποίο τρομοκρατεί τους πολίτες. Ένα καρτέλ ε, που δρά ανάμεσα στη Σλοβακία, Τσεχία και Λουξεμβούργο. Η περίπτωση, υπόθεση μάλλον 4075 κάθετος 2012 αφορά μια παρόμοια κατάσταση, μια παρόμοια υπόθεση σοβαρής επίθεσης κατά δικαιωμάτων των πολιτών και θέλουμε με τη δική μας ε, ε, αναφορά να ζητήσουμε να λυθεί αυτό το θέμα το οποίο ε, εξακολουθεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο εδώ και χρόνια γιατί οι Σλοβάκοι πολίτες κάνουν την πίστη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύντομη εκδοχή που έχετε λάβει έχει κατά κάποιο τρόπο παραμορφώσει ολόκληρη την αναφορά. Δεν ξέρω κατά πόσο την έχετε διαβάσει γιατί εμείς στο σημείωμα που λάβαμε ως απάντηση δεν απαντήσατε στην ουσία της αναφοράς αυτής. Αναφέρεται η Οδηγία 9546 και επίσης το γεγονός ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να επιλύσουν το συγκεκριμένο θέμα. Και στη δεύτερη απάντηση που λάβαμε μας είπατε για τα τέλη, τα τηλεοπτικά τέλη, ότι οι εθνικές αρχές είναι αρμόδιες για αυτά τα ζητήματα και αποφασίζουν για το τέλη που καταβάλουν οι πολίτες. Στην τρίτη απάντηση της Κομισιόν, η Κομισιόν δηλώνει ότι οποιοδήποτε πελάτης μπορεί να ακυρώσει τις υπηρεσίες εφόσον οι όροι και οι προϋποθέσεις παραβιαστούν. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να είμαι βέβαιος κατά πόσο η αντίδραση της Επιτροπής αυτής είναι παρεξήγηση ή αν ήταν θελημένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ακούσουμε και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα σας ξαναδώσουμε το λόγο στο τέλος για να, ε, να μας δώσετε καταληκτικές ε, παρατηρήσεις. Μα σας ε, έδωσα πέντε και μιλήσατε για επτά λεπτά. Στο τέλος μπορείτε να μιλήσετε για δύο λεπτά. Δεν έχουμε δύο λεπτά. Στο τέλος της συζήτησης μπορείτε να καταλήξετε. Στο τέλος της συζήτησης, όχι τώρα. Είχατε στη διάθεσή σας ε, πέντε λεπτά και ήδη μιλήσατε επί επτά. Μπορώ να συνεχίσω. Όχι. Μιλήσατε για επτά λεπτά. Αυτό σας είπα. Μιλήσατε για επτά λεπτά. Δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο τώρα. Ευνίκε Προκόπ από την ε, Επιτροπή για να μας ε, ε, μιλήσει και μετά, αφού και οι συνάδελφοι ε, λάβουν το λόγο, ε, θα σας δώσω το λόγο για δύο λεπτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ την Πρόεδρο από την DG Connect και την DG ε, just, τις δύο αυτές γενικές ε, διευθύνσεις, θα ήθελα να πω στον αναφέροντα ότι διαβάσαμε τη σύνοψη αλλά και το πλήρες κείμενο της αναφοράς από το οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο αναφέρθηκε ε, όπως είδαμε και με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής, ο αναφέρον θίγει πολλά ζητήματα. Το πρώτο αφορά την ελεύθερη πρόσβαση στις ε, τηλεοπτικές υπηρεσίες στη Σλοβακία. Επίσης, από τη στιγμή που ε, εξουσιοθωτήθηκε μία ιδιωτική εταιρεία να χειριστεί το όλο ζήτημα, υπήρξε μία μεγάλη χειραγώγηση και κερδοσκοπία κατά των χρηστών. Επίσης, ο αναφέρον λέει ότι το δικαίωμα στα προσωπικά δεδομένα παραβιάστηκε και οι σλοβαγικές αρχές ε, δεν επόπτευσαν το όλο καθεστώς. Η Επιτροπή με βάση τις ε, νομικές ε, αρχές που ισχύουν ανέλησε την κατάσταση με βάση τις αρμοδιότητες της για να αναλάβει δράση ενδεχομένως και ασχολήθηκε με τα λεγόμενα του αναφέροντα. Τώρα μιλώ σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και η συνάδελφος θα μιλήσει για τις τηλεοπτικές υπηρεσίες. Υπάρχει παραβίαση εάν γίνει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αν δεν έχουν τύχη επεξεργασίας, δεν ισχύει παραβίαση τότε. Ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τα στοιχεία του χρήστη και ισχύει η προστασία. Όμως στην αναφορά γίνεται λόγος για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, ε, δηλαδή που αφορούν τις προσωπικές σας πεπιθήσεις, τις θρησκευτικές σας ε, πεπιθήσεις, το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε ή τη σεξουαλική σας ζωή. Αυτά τα στοιχεία δεν χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα περίπτωση. Όταν γίνει επεξεργασία στοιχείων, ε, γίνεται επεξεργασία με βάση τις αρχές των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια της επεξεργασίας και δεν υπήρξε παραβίαση αυτών των δεδομένων. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο αναφέρον αναφέρθηκε σε ένα ισχυρισμό σε σχέση με παραβίαση δεδομένων μεταξύ φυσικού προσώπου και ιδιωτικής εταιρεία. Οι αρμόδιες αρχές είναι οι εθνικές αρχές. Γι' αυτό και η Επιτροπή στην ανακοίνωση ζήτησε από τον αναφέροντα να αναφερθεί στην Εθνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Εποπτείας για να ασχοληθεί με την ε, τρέχουσα προσφυγή. Αυτό σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ε, στη συνέχεια ο συνάδελφος ή η συνάδελφος θα μιλήσει για το άλλο σκέλος ε, της ερώτησης. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω και εγώ αναφερόμενοι στο θέμα αρμοδιότητας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση τηλεοπτικών σταθμών. Υπάρχει το πρωτόκολλο 29 για το σύστημα ε, δημόσιας μετάδοσης και το πρωτόκολλο αυτό αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη είναι ε, αρμόδια για τη χρηματοδότηση η οποία θα ε, διοχετεύεται σε οργανισμούς ε, τηλεπικοινωνιών. με τρόπο ο οποίος δεν θα πρέπει να δημιουργεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Είναι σαφές λοιπόν από το πρωτόκολλο αυτό ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τη διοργάνωση της ε, χρηματοδότησης και για τις ε, προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες της χρηματοδότησης αυτής. Ε, δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, όμως προς το παρόν και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε δεν βλέπουμε αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αναλάβει εποπτικό ρόλο ή έστω για να παρέμβει στην περίπτωση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη για σχόλιο. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε την πλευρά του κατά πόσο υπάρχει κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης. Εν προκειμένου ο αναφέρον είναι λήπτης υπηρεσιών και εδώ έχουμε μία υπηρεσία η οποία παρέχεται αντί ενός συγκεκριμένου ποσού. Μας είπε λοιπόν, από τα στοιχεία που έφερε τουλάχιστον, ότι αυτό το ποσό που απαιτείται προκειμένου να έχει, ελεύθερη προκειμένου να έχει πρόσβαση είναι αρκετά υψηλό. Δεύτερο, η εταιρεία αυτή είναι και η μοναδική η οποία παρέχει τις υπηρεσίες. Επομένως δεν έχει ανταγωνιστεί. Τρίτον, ότι σε περίπτωση που διακοπεί η παροχή της υπηρεσίας αναζητά αυτό με κάποιο τηλεφώνημα το οποίο είναι και ακριβώς ως ποσό που πληρώνει, αλλά και που από ό,τι λέει δεν βρίσκει και άκρη στα θέματα αυτά. Επομένω, θα έλεγα ότι η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει την περίπτωση να έχουμε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης και επομένως να έχουμε εδώ ένα μονοπόλιο το οποίο είναι ιδιωτικό μονοπόλιο και που ασκεί καταχρηστικά όλη τη δραστηριότητα η οποία έχει επίπτωση στον αναφέροντα ως λήπτη υπηρεσιών. Επομένως, εκτός από τα θέματα που τέθηκαν στις πλευρές που έθεσε η Κομισιόν, δηλαδή του πρωτοκόλλου 29 ή του ζητήματος της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ακόμη και αν πούμε ότι έχει δίκιο η Κομισιόν, που εγώ διαφωνώ σε κάποια θέματα που έθεσε η Κομισιόν, βλέπω ότι δεν έχει εξετάσει την κλασική περίπτωση ενός μονοπωλίου ιδιωτικού το οποίο παρέχει υπηρεσίες πάρα πολύ ακριβές και πλέον καταχράται τη δεσπόζουσα θέση την οποία έχει. Επομένως να, να δούμε αυτό από την σκοπιά πλέον του άρθρου περί ανταγωνισμού και μονοπωλίων παρότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και πολιτικά θέματα που έχουν σχέση με ενδεχόμενη ε, παραβίαση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αλλά αυτά πρέπει να μας δώσει περισσότερα στοιχεία ο αναφέρον όπως επίσης και το άρθρο 29 σε σχέση με την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ας το δούμε λοιπόν, παρότι πολιτικά το ξεκίνησε ο αναφέρον βάζοντας τα θέματα αυτά, ας το δούμε από την πλευρά την οικονομική, δηλαδή της εσωτερικής αγοράς και των μονοπωλιακών διαστάσεων που έχει συγκεκριμένη επιχείρηση. Ευχαριστώ. Άρα να γίνει παραδεκτή και να εξεταστεί παρακάτω η υπόθεση. Ευχαριστώ. Ο Πέτερ έχει το λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να κάνω μία σύσταση στον αναφέροντα, όπως είπε και η Κομισιόν, ε, να απευθυνθεί στις εθνικές αρχές, ε, στην Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Προτού φτάσουμε δηλαδή στον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή, υπάρχει μια εθνική αρμόδια αρχή και μια και πρόκειται για ε, δημόσια τηλεόραση, είναι εθνική αρμοδιότητα. Είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, γι' αυτό η διάσταση είναι εθνική. Ακούσαμε ότι ίσως είναι θέμα ευρωπαϊκής ε, νομοθεσίας ευρωπαϊκού δικαίου. Εγώ θα πρότεινα να περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει πρώτα σε εθνικό επίπεδο. Όταν ε, διευκρινιστεί το θέμα εκεί, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι ένα θέμα που αφορά τη δημόσια τηλεόραση, όπως είπα, και τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την δημόσια τηλεόραση και τη σύσταση αυτή. Ε, η προστασία δεδομένων είναι κάτι που πρέπει να εγγυηθούν τα κρατημέλη, η ουδετερότητα κτλ. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν βλέπω πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα εθνικό ζήτημα. Ε, προτείνω να κλείσουμε λοιπόν την αναφορά με την ε, αναφορά με τη σύσταση μάλλον να παραπεμφθεί στις εθνικές αρχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου, μια που έχουμε και Σλοβάκο αναφέροντα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία διαφορετικά σημεία της αναφοράς αυτής. Καταρχάς, είναι θέμα που ε, αφορά την Σλοβακία. Στη Σλοβακία υπάρχει αρχή προστασίας δεδομένων, προσωπικών δεδομένων. Είναι μια αρχή η οποία πρέπει να ασκεί τις αρμοδιότητές της και πιστεύω πως πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Έπειτα υπάρχει και η αντίστοιχη επιθεώρηση εργασίας στη Σλοβακία. Εμπορικό επιμελητήριο στη Σλοβακία. Θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε εκεί και να τους ρωτήσουμε εάν έχουν διαπιστώσει ε, παραβιάσεις ή κατάχρηση όπως ε, αναφέρεται στην αναφορά. Έπειτα. Μπορούμε να ζητήσουμε να μας δώσουν εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο απαιτούν ε, την καταβολή αυτών των τελών από τους ε, χρήστες. Έπειτα, όπως ε, ακούσαμε, η εταιρεία αυτή έχει έδρα στο Λουξεμβούργο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να επικοινωνήσουμε με τις αρχές του Λουξεμβούργου για να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Έπειτα, θα μπορούσαμε ίσως να ζητήσουμε μία γνωμοδότηση εδώ στο Κοινοβούλιο, ενδεχομένω από τις Επιτροπές Ήτρε ή Ίνκο για να ε, δώσουμε περισσότερο φως ε, στην ε, περίπτωση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. θα έχει ζητήσει κάποιο άλλος το λόγο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο πίσω στον κύριο Γιάννη Λούτεραν, τον αναφέροντα. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σχολιάσω ε, αυτά που είπε ο Σλοβάκος ε, Ευρωβουλευτής. Θα ήθελα να σας πω ότι τα βρίσκω πάρα πολύ θετικά, όμως δεν νομίζετε πως ε, αυτό είναι κάτι που το έχουμε κάνει. Δύο χρόνια πριν επικοινωνήσαμε με τις αρμόδιες αρχές, με το, με το Κοινοβούλιο της Σλοβακίας, με τον διαμεσολαβητή. Έχουν γίνει εκατοντάδες ε, υποβολές αναφορών ε, στο, στην Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Προωθήθηκε το ζήτημα στο εμπορικό επιμελητήριο, μετά προωθήθηκε το αντίστοιχο της Τσεχίας, μετά στο, στην αρχή τηλεπικοινωνίων της Τσεχίας, μετά επιβλήθηκε πρόστιμο 15 εκατομμυρίων ε, κορονών στην εταιρεία, όμως αυτό δεν φαίνεται πως είχε κάποιες ε, ε, θετικές επιπτώσεις, κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή η υπόθεση συνεχίζεται από το 2014 μέχρι σήμερα υπάρχουν χιλιάδες καταγγελίες που έχουν γίνει από τους ε, χρήστες των υπηρεσιών της εταιρεία αυτής και έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε και ό,τι προέβλεπε ο νόμος. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να συνειδητοποιήσετε ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Κάποιος κάπου χειραγωγεί ε, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Εσείς ως χρήστης πληρώνετε για κάποιες υπηρεσίες πληρώνεται την ε, εταιρεία για την μετάδοση προγράμματος και μετά η, η εταιρεία πληρώνεται από το κράτος και ταυτόχρονα ζητά και από τους χρήστες ξανά πληρωμή. Είναι μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση και η εντύπωση που έχω αποκομίσει είναι ότι δεν καταλαβαίνετε απόλυτα αυτό που θέλω να πω. Αυτή η περίπτωση αφορά εκατοντάδες, χιλιάδες οικογένειες. Ε, ξέρετε, λαμβάνουν επιστολή τα νοικοκυριά και στην επιστολή ε, αναγράφεται ότι αν δεν πληρώσετε τόσα και τόσα τέλη δεν θα έχετε τηλεόραση. Θα σας κόψουμε τη μετάδοση. Θα σας ακυρώσουμε τον αναμεταδότη. Το 51% ε, των ραδιομεταδόσεων στη Σλοβακία όταν ιδιωτικοποιήθηκαν πήγε στην ε, Deutsche Telekom, ξέρετε. Είναι φαύλος κύκλος, δεν βρίσκουμε λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ που σας διακόπτω, λέει η Πρόεδρος, στη μέση της πρότασής σας, αλλά ε, χρησιμοποιήσατε περισσότερο χρόνο από αυτόν που σας είχε δοθεί. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που ε, σταματήσατε και θα προσπαθήσω να συνοψίσω τις προτάσεις που έχουν γίνει από τους συναδέλφους. Καταρχάς, θεωρώ ότι και ο κύριος Εμεριάς και ο κύριος Ζάκη θέλουν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπατε. Θα την κρατήσουμε λοιπόν ανοιχτή. Και επίσης, Θέλουμε να πούμε σε εσά, κύριε Λούτεραν, ότι οι ανησυχίε σα ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από αυτήν την Επιτροπή. Και όσον αφορά το θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορούμε να συντάξουμε μία επιστολή για την αρχή εποπτείας προσωπικών δεδομένων του Λουξεμβούργου και την ε, αντίστοιχη αρχή στην Σλοβακία και να τους ζητήσουμε μία απάντηση. Τώρα, σε σχέση με τους όρους του, των συμβολέων, θα μπορούσαμε να παραπέμψουμε την υπόθεση στις αρχές ε, της Σλοβακίας, στο εμπορικό επιμελητήριο της Σλοβακίας και ε, θα μπορούσαμε να παραπέμψουμε την αναφορά στις επιτροπές Ήτρε και Ίνκο, διότι είναι οι αρμόδιες επιτροπές για ε, τέτοιες περιπτώσεις συμβολέων και κρατώντας ανοιχτή την αναφορά θα επανέλθουμε. Εσείς τι άποψη έχετε κύριε Μαριά. Να ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους ε, όρους του συμβολέου, τι γίνεται εκεί. Διότι υπάρχει, υπάρχει εδώ περίπτωση κατάχρησης εξουσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα μπορούσε να εξετάσει το θέμα αυτό. Ναι, είναι όμως αρμοδιότητα των κρατών μελών για να ορίσουν τις ε, λεπτομέρειες σχετικά με τη χρηματοδότηση της ε, δημόσιας τηλεόρασης. Όχι, όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι στο άρθρο 86 και την θέση εξουσίας. Είναι κάτι άλλο. Ο αναφέρον εδώ δέχεται υπηρεσίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ υπάρχει περίπτωση μονοπωλίου που κάνει κατάχρηση εξουσίας. Και αυτή η περίπτωση ενδεχομένως να ε, υπάγεται και στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα έπρεπε να εξετάσει το ζήτημα και αν διαπιστωθεί όντως τέτοια περίπτωση κατάχρησης να προχωρήσει ε, σε περαιτέρω εξέταση εγώ το εξετάζω από την εμπορική και οικονομική του πτυχή και όχι τόσο από την ε, πολιτική του διάσταση ή ε, για τα δικαιώματα των ε, πολιτών στην πληροφορία από τις εθνικές αρχές. Είναι, είναι, είναι κάτι τελείως οικονομικό, εμπορικό το ζήτημα, έτσι όπως το εξετάζω. Μάλιστα. Θα στείλουμε λοιπόν την αναφορά στην Επιτροπή, όπως το είπατε, και μαζί με τα υπόλοιπα που έχουν ήδη προταθεί και σας ανέφερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω ξανά τον κύριο Λούτεραν. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας και αναφέρατε το θέμα σας. Δυστυχώς θα πρέπει να εγκαταλείψω την αίθουσα τώρα και ο Παλτσάκη θα αναλάβει καθήκοντα Προέδρου. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Και θα δω τους υπόλοιπους από εσάς αύριο το πρωί. Uh, Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Το επόμενο θέμα, η επόμενη αφορά 2338 του 2013 από τη, από τη Μαρία Ναβάρο Διέγκο από πλευράς του ε, Habitat. Εδώ έχουμε δύο αναφέροντες από την Ισπανία. Έχετε το λόγο. 5 με 6 λεπτά το πολύ. Έχετε το λόγο. Εμείς πολίτες της Ένωσης θα θέλαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου ε, κυριαρχεί η φωνή του λαού να μπορέσετε να επανορθώσετε την κατάσταση σε σχέση με τις αδικίες της ισπανικής κυβέρνησης δεν δόθηκε επιδότηση ε, στέγης σε χιλιάδες ε, πολίτες της Ισπανίας όπως προβλεπόταν. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η κοινότητα της Βαλένθια, η τοπική κυβέρνηση καταχράστηκε την ε, δεσπόζουσα θέση της και δεν χορήγησε τις επιδοτήσεις σε χιλιάδες οικογένειες σε περίπτωση κάλυψης των αναγκών στον τομέα της στέγασης. Πρόκειται για 300.000. Αυτές είναι οι οικογένειες που πλήττονται και αναδρομικά θα έπρεπε η κυβέρνηση της Ισπανίας να καλύψει αυτές τις οικογένειες. Πρόκειται για οι οικογένειες που μέσα στα πλαίσια της ε, φούσκας των ακινήτων μπόρεσαν να αποκτήσουν στέγη στην ε, οποία τώρα δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Αυτές οι οικογένειες θα πρέπει να καλύψουν το κόστος των ε, υποθηκών τους καταβάλλοντας πολύ περισσότερα χρήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με βάση τη γενικευμένη οικονομική κρίση. Η κυβέρνηση της Ισπανίας δυστυχώς παραβίασε τις υποχρεώσεις της, αθέτησε τις υποχρεώσεις της με βάση τον νόμο περί κοινωνικής στέγης και γι' αυτό δεν τήρησε τις συνθήκες περί ασφάλειας δικαίου. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αυτή την κατάσταση, κατάσταση τη στιγμή που κατέφυγαν σε δανειοδότηση οι κάτοικοι αυτοί, στην οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν λόγω της αλλαγής της κατάστασης. Επίσης, επικράτησε νομικό χάος γιατί δεν ευεργετήθηκαν οι ίδιοι και παράλληλα η κυβέρνηση, αυτόνομη κυβέρνηση της Βαλένθια δεν ε, μπόρεσε παρά να υπερβεί τις 280.000 χρέους αυτών των πολιτών. Μεταξύ 5 και 12 η Generalitat της ε, Βαλένθια χειρίστηκε διαφορετικά την ε, επιδότηση δανείων και γι' αυτό στο τέλος ε, καρπόθηκαν τα κέρδη οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Και γι' αυτό ακριβώς δεν λήφθησαν υπόψη ανάγκες 6.000 οικογενειών και δυστυχώς δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην ε, κάλυψη των αναγκών τους. Εάν λάβουμε υπόψη τα έξοδα αυτά, ζήτησαν οι δικαιούχοι ε, αρρωγή η οποία δυστυχώς έτυχε αυθαίρετης αντιμετώπισης από τις αρχές. Το 2014 ε, χρειάστηκε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Κερδίσαμε σε 15 υποθέσεις και έτσι ορίστηκε ένα χρονοδιάγραμμα καταβολής ε, δαπάνων. Μιλάμε για για 60 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την ε, Ισπανική κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις επιδοτήσεις στέγης και να αναθεωρήσει το καθεστώς επιτοκίων που ισχύουν. Επίσης, η Ισπανική κυβέρνηση και η κυβέρνηση της Βαλένθια θα πρέπει να αναθεωρήσει το καθεστώς και να δούμε και ποιες πολιτικές ευθύνες απορρέουν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ε, ε και εκπρόσωπο από την Επιτροπή που προέρχεται ίσως και από την περιοχή της ε, Βαλένθια. Ευχαριστώ πολύ. Καθώς μιλάμε, ε, η διευθύντριά μας είναι ακόμα στο δρόμο για αυτή την συνεδρίαση γιατί έφτασε λίγο αργοπορημένα με αυτή την πτήση και δεν θα τα καταφέρει για να μιλήσει άμεσα. Εξ ονόματος λοιπόν της ε, τοπικής κυβέρνησης της αυτόνομης περιοχής της Βαλένσια. σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε να συζητήσουμε αυτό το θέμα όλοι μαζί. Το πρόβλημα της μη καταβολής των στεγαστικών επιδομάτων που προέκυψε από, μια, ένα, διάταγμα, ε, προέκυψε από ένα διάταγμα της ε, κυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος το 2012. Η εθνική κυβέρνηση ακύρωσε επιδοτήσεις που ήδη είχαν δοθεί σε ισπανικές οικογένειες για την αγορά πρώτης κατοικίας σύμφωνα με το πλάνο ε, πρώτης κατοικίας. Επίση υπήρξαν διαφορετικέ ερμηνείε στην νομοθεσία από το αρμόδιο Υπουργείο. Για να εφαρμοστεί αυτό η νομοθεσία του 2012 μειώθηκε βία και κάθετα ο προπολογισμό. Είχαν προβλεφθεί 120 εκατομμύρια το 2009 και κατέβηκαν στα, μόνο στα 11 εκατομμύρια το 2014 αυτή η προβλεπόμενη επιδότηση. Ο αντίκτυπο ήταν τεράστιο. 500.000 δικαιούχοι επηρεάστηκαν. Το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων πιστοποίηση που ήδη είχα χορηγηθεί ήταν 250 εκατομμύρια ευρώ. Ευτυχώς Μπορούμε να πούμε ότι η σημερινή κατάσταση, σήμερα η κατάσταση είναι διαφορετική. Πέρυσι η περιφέρεια της Βαλένθια επέλεξε νέα κυβέρνηση αλλαγής με πιο καθολική κοινωνική ατζέντα που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο. Από τον Ιούλιο αυτή η νέα κυβέρνηση αντέδρασε μέσω στο νέο, σε αυτό το πρόβλημα των μη καταβεβλημένων επιδοτήσεων και στις πρώτους μήνες ε, ε, ε, λειτουργίας της ε, ρύθμισε ε, ένα σχέδιο πληρωμών για όλες τις μη καταβεβλημένες επιδοτήσεις. Από τα 250 εκατομμύρια έχουν καταβληθεί ήδη 210 εκατομμύρια και παραμένουν ακόμα 40 εκατομμύρια για τους ανθρώπους που δεν έχουν επιδοτηθεί τα, η καταβολή των τελευταίων 40 εκατομμυρίων θα, θα συμπληρώσει ε, και θα ολοκληρώσει τα ποσά προς όφελος όλων αυτών των οικογενειών που επηρεάστηκαν από αυτή την κατάσταση και αυτό είναι το μήνυμα της ε, περιφερειακής κυβέρνησης της Βαλένθια. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να ρωτήσω ποια είναι η θέση της Επιτροπής. Κυρία Λάουρα Αγγεμαναρελάνο από την DG Regio. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ και συνάδελφος Στέφανη Γολφχάρταν, είμαστε παρούσες από την DG Radio και έχουμε έρθει για να διευκρινίσουμε κάποιες νομικές πτυχές σε αυτήν την ε, αναφορά τη απουσία της DG Justice που δεν μπορούσε να είναι εδώ. Καταρχάς με χαρά ακούω η κατάσταση σιγά σιγά βελτιώνεται. Ήδη πολύ καλά είναι τα νέα. Η Κομισιόν ανησυχεί πολύ για την επίλυση αυτής της, αυτού του προβλήματος που περιλαμβάνει ένας, και επηρεάζει ένα σημαντικό στοιχείο της ευημερία των Ευρωπαίων, δηλαδή πρόσβαση στη στέγαση, κοινωνική ένα μέτρο για την καταπολέμηση της στόχης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πολύ σημαντικό για χώρες όπως η Ισπανία που χτυπήθηκαν πολύ έντονα από την οικονομική κρίση και έχουν ε, ε, οδηγηθεί σε αυξημένα επίπεδα κοινωνικού αποκλεισμού. Η πολιτική στέγαση είναι ευθύνη των κρατών μελών. Ωστόσο, η πολιτική συνοχή παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό το τομέα, ιδιαίτερα μέσω τη στήριξη στι βελτιώσει για ε, επάρκεια στην ενέργεια και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Επίση, στηρίζουμε την κατασκευή νέων καταλήμματων υπέρ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν συμπληρωματικέ δράσει στον τομέα τη παιδεία, τη υγεία και της υγειονομικής περίθαλψης. Εδώ όμως δεν έχουμε ε, ε, κοινωνικό ταμείο, οπότε η Κομισιόν δεν μπορεί δυστυχώς να παρέμβει. Αυτή τη στιγμή η Στεφανή Ρελού θα πάρει το λόγο για να εξηγήσει με περισσότερες λεπτομέρειες αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ε, ήθελα να σας δώσω κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες ε, για την νομική φύση αυτής της αναφοράς. Ε, ιδιαίτερα αυτό το άρθρο 34 που αναγνωρίζει δικαιώματα για βοήθεια στη στέγαση. Εγώ, όπως είπε και η συνάδελφος, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εδώ. Πρόκειται για εθνικές επιδοτήσεις και όπως ορίζει το άρθρο 51 του χάρτη, ο Χάρτη ε, είναι εφαρμόσιμο στα κράτη-μέλη μόνο όταν εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οπότε είχαμε κάποια δυσκολία να κάνουμε τη σύνδεση ανάμεσα στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και το Εθνικό Σχέδιο Επιδοτήσεων. Οπότε σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση η Κομισιόν δεν μπορεί να παρέμβει όσον αφορά τι επιδοτήσει. Σα ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Από ό,τι κατάλαβα, η ε, ε, περιφερειακή κυβέρνηση είναι έτοιμη να λύσει το πρόβλημα. Εγώ σας είπα ότι δεν είμαι όμως υπεύθυνο για αυτό το θέμα. Είμαι εδώ εξ ονόματος της περιφέρειας της Βαλένθια και από τις πληροφορίες που έλαβα φαίνεται πως 200... 35 εκατομμύρια έχουν ήδη πληρωθεί και καταβληθεί και άλλα 15 πρόκειται να καταβληθούν σύντομα. Υπάρχει δηλαδή η βούληση και έχει ήδη γίνει ένα σχέδιο για την καταβολή των επιδοτήσεων. Ξεκινάμε με την κυρία Ροντρίγκε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, καταρχάς να καλωσορίσω, αν και δυστυχώς ήρθαν για αυτή την υπόθεση, η Ένωση σύνδεσμο μάλλον των ε, δικαιούχων ε, για τις τα μη καταβληθέντα επιδόματα. Εγώ καταλαβαίνω τα όσα είπε η Κομισιόν, όσα είπε η Κομισιόν είναι σωστά, αν και... Είναι δέσμευση αυτής της Επιτροπής να διευκολύνει προγράμματα που στόχο έχουν την πρόσβαση στην στέγαση. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν κοινοτικά κονδύλια. Όμω θέλω να ξέρω τι έχει γίνει σε σχέση με τι αρχέ τη νομική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτή την ανάλυση για μήπω και βρεθεί κάποια λύση. Σε τι αναφέρομαι. Όταν ένα κράτο μέλο χρησιμοποιώντα ε, το δικαίωμα και τι αρμοδιότητέ του αποφασίζει με βάση κάποιου κανόνε να θεσπίσει ορίσει όρους υπό τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να έχουν πρόσβαση. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι Εάν σεβαστούμε τις αρχές της ε, νομικής βεβαιότητας και της ε, νομικής εμπιστοσύνης είναι να αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στα μέσα της, του παιχνιδιού. Και αυτό συνέβη με την κυβέρνηση της Ισπανίας. Γιατί κάποιοι όροι που πάντοτε ανανεώνονταν αυτόματα ε, μετά από πολλά χρόνια σχεδίων στέγασης της Ισπανίας ανανεώνονταν οι ίδιοι, οι ίδιοι όροι και επιδοτούνταν τα δάνεια. Λοιπόν, πάντα ήταν έτσι και ποτέ δεν ε, ε, προειδοποιήθηκε κανείς ότι επρόκειτο να αλλάξει κάτι. Το αποτέλεσμα ήταν λοιπόν ότι εφόσον δεν παρατάθηκαν οι ίδιοι όροι και συνθήκες ε, τη στιγμή του ξεσπάσματος αυτής της τόσο έντονης και βίαιης οικονομικής κρίσης ε, που χτύπησε την Ισπανία και ιδιαίτερα στη Βαλένσια μέχρι και που έχασαν τελείως τη δουλειά τους πολλές οικογένειες. Πολλές οικογένειες λοιπόν που καλή την πίστη είχαν πάρει δάνεια και λόγω της νομικής βεβαιότητας που δίνει ένα ολόκληρο κράτος είδαν ότι άλλα άλλαξαν οι παιχνιδιού και δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τι υποχρεώσει του. Και πολλοί χρειάστηκε να φύγουν από τα σπίτια του. Ε, ε, ε, γίνανε εξώσει δηλαδή. Από αυτή τις βάσεις λοιπόν θα ήθελα να διαβιβάσω στην Κομισιόν και στην Επιτροπή των Αναφορών αυτή την κατάσταση. Σε σχέση τώρα με την ε, περιφερειακή κυβέρνηση, η αλλαγή της κυβέρνησης είναι επίσης μια αλλαγή ε, κάθετη και υπάρχει ένα θέμα πολιτικής βούλησης και σε μια στιγμή όπου βρεθήκαμε με άδεια τα ταμεία λόγω της πολιτικής κατασπατάλησης και διασπάθησης χρήματος εντός της κυβέρνησης, της αναλήφθη μια υπόσχεση ε, και ένα χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των επιδομάτων αυτών παραπάνω τώρα. Θα πρέπει να καθοριστούν ε, τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή τη συμπεριφορά και όσον αφορά την έρευνα να δούμε αν ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα τα οποία είναι σκόπιμα ώστε να καταλογιστούν οι ευθύνες. Με όλη τη στήριξη λοιπόν της σημερινής ε, ε, ε, κυβέρνησης της Βαλένθια αλλά και των βουλευτών από τη Βαλένθια που είμαστε εδώ παρόντες ελπίζουμε ότι θα λυθεί πλέον το πρόβλημα. Η κυρία Αλμπιόλ καταρχήν να καλωσορίσω την Ένωση των Εκπροσώπων και θα ήθελα να πω ότι έχουν δώσει μεγάλη μάχη κατά τη διάρκεια πολλών ε, χρόνων και πολλές φορές ζήτησαν δικαίωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να τους δώσουμε ικανοποιητική απάντηση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η κατοικία είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα όπως ορίζει και ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων και κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων. Κάτι το οποίο δεν τηρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ζούμε σε μία κρίση της κατοικίας με εκατομμύρια ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ε, λιτότητας και περικοπών που ε, ζει η Ιρλανδία η Ελλάδα και η Ισπανία μεταξύ άλλων. Για δεκαετίες η κατοικία θεωρήθηκε όχι δικαίωμα αλλά δικαίωμα για την κερδοσκοπία και αυτό σε σχέση με την ε, δημόσια κατοικία και την κατοικία που αφήσαμε στα χέρια της αγοράς. Υπάρχουν 500.000 άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στην ε, κατοικία στην Ισπανία. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπήρξε δημόσια πολιτική για την κατοικία και αφέθηκαν τα πάντα στα χέρια των ε, κερδοσκόπων. Μιλάμε για ένα 1% ε, τη δικαιώματος στην κατοικία, ενώ στην Ισπαν... στη γαλλια αντιστοιχω αντιστοίχως υπάρχει ένα 17-18% και 18% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν ότι μειώθηκε ο κρατικός ε, υπολογισμό μεταξύ 2005 και 2016. Αυτό σε σχέση με την δημόσια προστασία της κατοικίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αναφέροντες έχουν πληγεί γιατί δεν υπάρχει πολιτική θέληση. Υπάρχει λοιπόν η καταγγελία έναντι του κράτους διότι το κράτος αναδρομικά ε, αφαίρεσε το δικαίωμα προστασίας των ενυπόθηκων δανείων και ιδιαίτερα στη Βαλένσια διότι η αυτόνομη κυβέρνηση δεν κάλυψε τις επιδοτήσεις που προβλέπονταν για τις οικογένειες, γιατί επρόκειτο για εκπροσώπους της κυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος που δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους. Μιλάμε για χιλιάδες οικογένειες που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα ενυπόθηκα δάνειά τους. Και φυσικά ε, τώρα φαίνεται ότι με την αλλαγή κυβέρνησης επιλύεται το θέμα. Αυτό αφορά την περιοχή της ε, Βαλένσια. Δεν έχει επιληθεί το θέμα σε εθνικό επίπεδο. Μιλάμε για θέτηση λοιπόν του κοινοτικού δικαίου ως προς το δικαίωμα της ε, κατοικίας δυνάμει του άρθρου 31,4 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και από την άλλη πλευρά ε, δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου. 50.000 οικογένειες επλήγησαν διότι αναδρομικά τους αφαιρέθηκε αυτή η επιδότηση για να μειωθεί το δημόσιο χρέος και το δημόσιο έλλειμμα. Άρα, μη τηρώντας αυτά τα δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προώθησε την ιδιωτικοποίηση και την πολιτική της λιτότητας, καθώς και τη μείωση των ε, κοινωνικών πολιτικών υπέρ της κατοικίας. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ανταγωνισμός μόνο όταν υπάρχουν συμφέροντα η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σήμερα λέει ότι η πολιτική κατοικίας θα πρέπει να ισχύει είναι η ίδια η οποία επέβαλε στην Ελλάδα αλλαγή των νόμων έτσι ώστε να υπάρξουν εξώσεις από την πρώτη κατοικία. Άρα άλλα λέμε στην περίπτωση της Ελλάδας για τις ε, εξώσεις από την πρώτη κατοικία και από την άλλη πλευρά για την περίπτωση Βαλένσια τι μας λέει η Επιτροπή ότι δεν έχει αρμοδιότητες. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Η Επιτροπή αναφορών θα πρέπει να υποστηρίξει τους αναφέροντες και θα πρέπει να αποσταλεί μια επιστολή προς την κυβέρνηση μιλώντας ε, για εξαίρεση στην περίπτωση της αναδρομικής ε, αυθαίρετης μη ισχύω της πολιτικής επιδοτήσεων και αυτά τα χρήματα που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δεν δόθηκαν στους ε, τελικούς δικαιούχους δεν καταβλήθηκαν. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στη δεύτερη καταγγελία ως προς την αθέτηση του κοινοτικού δικαίου και την ανασφάλεια δικαίου με την άρση των επιδοτήσεων. Η Επιτροπή απάντησε σε ένα σκέλος, αλλά δεν μίλησε για την ανασφάλεια δικαίου σε σχέση με τους καταναλωτές. Καταλαβαίνω ότι είναι μία συζήτηση που αφορά το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία και θα ήταν σκόπιμο σε αυτή την Επιτροπή να γίνει μία συζήτηση για το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία και να προβάλλουμε μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για το δικαίωμα στην κατοικία σε ολόκληρη την Ευρώπη και να υποβάλουμε και προφορική ερώτηση για την συνέχεια που θα δοθεί υπό το φως της, του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σε σχέση με το δικαίωμα στην κατοικία. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες που είναι εδώ γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε με το θέμα αυτό. Ε, ξέρουμε ότι είχαν να ζήσουν αυτό το γολγοθά και είχαν να αντιμετωπίσουν και το συνταγματικό δικαστήριο. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για την κυβέρνηση της ε, Ισπανίας, αλλά για την υποχρέωση των κοινοτικών θεσμικών οργάνων να είναι θεματοφύλακες του χάρτη των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα σας υποστηρίξουμε οι Ισπανοί, αλλά και όλοι οι ευρωβουλευτές γιατί θα πρέπει να τηρούμε το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων γιατί πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με την ερμηνεία του άρθρου 51 κάτι το οποίο μας απασχόλησε γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το νομοθετικό κόρπους που αφορά και τους αναφέροντας. Εδώ πρόκειται για ένα πολιτικό ζήτημα. Θα θέλαμε ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς να αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα αύριο, αλλά θα ήθελα να πω ότι πράγματι υπάρχει ένα νομικό ζήτημα και η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα γιατί θα πρέπει να δει πώς προβάλλει την ερμηνεία του όλου ζητήματος. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους, τους πιο ευάλωτους. Αυτό πρέπει να κάνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως και η ισπανική κυβέρνηση και ε, δεν μπορούμε να πλήξουμε περαιτέρω αυτούς που είχαν δείξει εμπιστοσύνη στη κυβέρνηση και τις ε, πολιτικές της. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν το κόστος της ε, πρώτης κατοικίας, πώς διαμορφώνεται. Νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή το εξής. Να μας πείτε γιατί τα επιτόκια που ίσχυσαν ε, αρχικά για την κατοικία εξελίχθηκαν ε, με τον τρόπο που εξελίχθηκαν. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής, γιατί αυτό δεν έχει σχέση αποκλειστικά ε, με θέματα αρμοδιοτήτων για την πρώτη κατοικία. Το θέμα των επιτοκίων αφορά την Κομισιόν και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί η προστατευόμενη κατοικία βρίσκεται πάνω από συμφέροντα ε, τύπου Euribor. Νομίζω ότι αυτό το θέμα μας απασχόλησε και την ε, προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο μέσα στα πλαίσια της ε, καταπολέμησης της φτώχειας. Η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι θεμελιώδες δικαίωμα, το δικαίωμα της στέγης και θα πρέπει να υπάρχει σωστή πρόσβαση στην πρώτη κατοικία με ε, ηλεκτροδότηση και όλα τα βασικά δικαιώματα. Αυτό αφορά και την απασχόληση, την αξιοπρεπή απασχόληση και άλλους τομείς. Θα πρέπει να δούμε πώς ορίζουν τα κράτη-μέλη τις κοινωνικές επενδύσεις μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης 2020. Θα ήθελα να τονίσω ότι εδώ θα έπρεπε οι Ευρωπαίοι πολίτες να ασχοληθούν με την μία θέτηση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και να προασπίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα ήθελα η Επιτροπή να μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το αίτημα σε σχέση με το θέμα του Euribor και των επιτοκίων κατοικίας. Η κυρία Φεραγκούτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω την Ένωση των Πληγέντων από τα ενυπόθηκα δάνεια και θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς το Λαϊκό Κόμμα και η κυβέρνηση δεν αντιμετώπισαν σωστά το ζήτημα και τώρα που ήρθε η αριστερά άλλαξαν τα πράγματα. Τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε σε καλούς και κακούς και στην ουσία να χειραγωγήσουμε αυτή την επιτροπή υπέρ μίας ή άλλης κυβέρνησης δεν θα υπηρετούσαμε ούτε την Επιτροπή μας, ούτε την πολιτική. Όπως ξέρετε, η Ισπανία διήνυσε μια μεγάλη κρίση που άρχισε το 2012. Γι' αυτό και το συνταγματικό δικαστήριο και τα εθνικά δικαστήρια αποφάνθηκαν επί των επιδοτήσεων οι επιδοτήσεις αυτές δεν ήταν ε, μόνιμο δικαίωμα. Γι' αυτό ε, θελήσαμε να βοηθήσουμε τους ε, ευάλωτους και ιδιαίτερα εκείνους που δεν μπορούσαν να καταβάλουν ούτε το ενίκιό τους. Όμως κρίθηκε ότι δεν μπορούσαν να παραταθούν αυτές οι επιδοτήσεις και το Συνταγματικό Δικαστήριο καθώς και τα εθνικά το 2015 αποφάνθηκαν έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση όπως ίσχυε μετά το 2012. Χρειάστηκε λοιπόν ερμηνεία του άρθρου 35 για να βοηθήσουμε τις τοπικές αρχές. Μιλάμε για ένα μεγάλο χρέος 450 εκατομμυρίων, το οποίο κληρονομήσαμε από τους σοσιαλιστές και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Δεν υπήρξε καμία παρατυπία και πάντα λειτουργήσαμε με καλή πίστη. Η αυτόνομη κοινότητα της Βαλένσια είχε περίπου 200 ε, εκπροσώπους από πλευράς ε, περιφερειών στην εθνική κυβέρνηση. Ε, θα πρέπει να είμαστε αρκετά ουδέτεροι, δεν είμαστε καλοί και κακοί. Υπήρχε ένα ποσό 250 εκατομμυρίων που εκρεμούσε ένα μεγάλο χρέος της Βαλένθια, το οποίο δεν μπόρεσε να καλυφθεί και όταν ψήφισε το Λαϊκό Κόμμα τότε άρχισαν οι πληρωμές. Ήδη από το Δεκέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιούλιο του 2015 καλύφθηκαν 100, τα 150 εκατομμύρια και μετά καταβλήθηκε το υπόλοιπο. Ε, ο καθένας έκανε αυτό που μπόρεσε. Δεν υπάρχουν καλοί ή κακοί και το Λαϊκό κόμμα και όλοι προσπάθησαν να καλύψουν τα 250 εκατομμύρια που εκκρεμούσαν. Τώρα θα πρέπει να καταβληθούν 40 ή γύρω στα 30 εκατομμύρια που υπολείπονται. Ζήσαμε μία πολύ δύσκολη κατάσταση που δεν αφορούσε μόνο την Βαλένθια αλλά ολόκληρη την Ισπανία. Κάντε ό,τι διαβουλεύσεις θέλετε όπως είπε και η κυρία Βεφέρα, αλλά θα πρέπει να θέτουμε τα πράγματα στη σωστή του βάση, γιατί θα πρέπει να υπάρχει πολιτισμός και αξιοπρέπεια. Όλα τα πολιτικά κόμματα είμαστε, δείχνουμε μεγάλη ευαισθησία σε όλες τις ευάλωτες κατηγορίες. Η κυρία Βολέρο. την ώρα. Δεν πρόκειται για το θέμα κατά πόσο το ΕΛΚ είναι καλό ή κακό. Μιλάμε για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε, όπως είπε και η Ένωση, πώς έχουν τα πράγματα. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την περίπτωση της Βαλένθια και της Ισπανίας, όπου δυστυχώς επλήγησαν οι συνθήκες πρόσβασης σε μια αξιοπρεπή κατοικία. Όπως είπε και η συνάδελφος, δεν μπορεί να επικρατούν τα συμφέροντα του Γιούριμπορ και όχι των ανθρώπων. Ε, γνωρίσαμε μία ε, ιδιάζουσα κατάσταση στην Ισπανία και το ζήτημα είναι να δούμε και την περίπτωση της Αστούριας όπου ε, χτίστηκε ένα, ένα μεγάλο συγκρότημα όπου μπορέσαμε να χορηγήσουμε 45.000 κατοικίες σε πολίτες. Στις Αστούριας είδαμε ένα παράδειγμα και εκεί δεν γίνανε εξώσεις από την ε, κατοικία από την, και ειδικά από την πρώτη κατοικία. Πολλοί λένε ότι το θέμα αυτό δεν αφορά ε, ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία είναι ένας από τους τρόπους για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και την κοινωνική αδικία. Και πιστεύω ότι το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία είναι ένα θέμα που επλήγει στην Ισπανία από την κερδοσκοπία, από τις ε, περικοπές και από άδικους νόμους. Όπως ξέρετε και το ΔΕΚ καταδίκασε την Ισπανία και καταγγέλθηκε το ζήτημα αυτό και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς τις ε, εξώσεις και τα ενυπόθηκα ε, δάνεια. Και μέσα στα πλαίσια του δημοσίου συνήγορου ε, δόθηκαν νέες προθεσμίες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Φυσικά δεν τηρήθηκε ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα ήθελα να υποβάλουμε μια προφορική ερώτηση και στην κυρία Τίσεν που ασχολείται με την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα για να μας δώσει μια σαφή απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και ίσως υπάρχει και καλή θέληση από τις Ισπανικές αρχές να επιλύσουν αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό θα ήθελα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να ε, αποστείλουμε μία επιστολή στην κυβέρνηση της Βαλένθια για να δούμε πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση και όταν λάβουμε απάντηση τότε θα κλείσουμε την αναφορά με βάση το κατά πόσο έχουν ανταποκριθεί. Μπορείτε να το δεχτείτε. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, έχετε το λόγο. Θα ήθελα απλώς να προσθέσω σε σχέση με μία περαιτέρω επεξήγηση της Επιτροπής σε σχέση με το Euribor να γίνει εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών. Δεν αντιτίθεμαι εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα της Επιτροπής σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ποια είναι η θέση σας γιατί φαίνεται ότι αυτό είναι εσωτερικό ζήτημα της Ισπανίας. Δεν μπορώ να απαντήσω. Μπορείτε να το υποβάλλετε στην Επιτροπή, αλλά δεν ξέρω ποια γενική διεύθυνση θα ήταν αρμόδια για να απαντήσει ένα τέτοιο ερώτημα. Όχι η Γενική Διεύθυνση Ρίγκιο, αυτό είναι σίγουρο. Ίσως η Γενική Διεύθυνση Just θα μπορούσε να απαντήσει σε σχέση με θέματα ε, ασφάλειας δικαίου και νόμιμης εμπιστοσύνης που ίσως δεν καλύφθηκαν. Ίσως η Γενική Διεύθυνση Justice να μπορέσει να σας δώσει απαντήσεις. Τώρα, γιατί τα επιτόκια ανέβηκαν πάνω από το Euribor, δεν ξέρω, εσείς θα κρίνετε κατά πόσο πρέπει να θίξετε αυτό το θέμα με την Επιτροπή. Άρα το αίτημά σας είναι ακριβώς αυτό. Δεν είμαι απολύτως σίγουρη ποια γενική διεύθυνση πρέπει να απαντήσει, αλλά εδώ υποβλήθηκαν ερωτήματα ε, που ίσως και η κυρία Τίσεν, ε, η Επίτροπος, θα μπορούσε να απαντήσει. Ίσως η Επιτροπή θα απαντήσει μέχρι ποιου σημείου θα πρέπει να απαντήσει. Εμείς θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Επίτροπη, όχι σε μια συγκεκριμένη γενική διεύθυνση εξ ονόματος της ε, δικής μας Επιτροπής. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Σας συστήνω λοιπόν να δείτε ποια γενική διεύθυνση είναι υπεύθυνη και θα προετοιμάσουμε μία επιστολή. Το δέχεστε? Εσείς αποφασίστε ως Προεδρείο, αλλά δεν αποστέλουμε τις επιστολές σε μια συγκεκριμένη γενική διεύθυνση, αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσατε να το επαληθεύσετε αυτό ή πριν ή μετά. Εντάξει. Θα αποστείλουμε μία επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Το πιο σημαντικό ζήτημα που έφυξαν οι αναφέροντες είναι η, κατάργηση του αναδρομικού αυτού χαρακτήρα άρσης των επιδοτήσεων και να τους δώσουμε μία απάντηση. Θα ήθελα να γίνει και κάποια σύσταση από την ε, Επιτροπή ζητώντας εξαίρεση από την αναστολή της επιδότησης. Ίσως θα μπορούσαμε να αποστείλουμε αυτή την ε, επιστολή ε, κάνοντας ορισμένες παρενέσεις προς την Ισπανική κυβέρνηση και επίσης μετά από τη συζήτηση θα ήταν σκόπιμο να ακούσουμε και τους αναφέροντες. Με τη λήξη της συζήτησης. Ναι, αλλά αν κατάλαβα καλά, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της ε, κεντρικής κυβέρνησης αλλά της ε, περιφερειακής. Θα αποστείλουμε δηλαδή την επιστολή στην περιφερειακή κυβέρνηση. Το θέμα της επιδότησης αφορά την κυβέρνηση, την κεντρική κυβέρνηση. Υπάρχουν δύο θέματα. Το θέμα της επιδότησης που αφορά το κράτος και την μη καταβολή των επιδοτήσεων που αφορά τη Βαλένθια το οποίο φαίνεται ότι επιλύεται. Όμως το θέμα σε κρατικό επίπεδο δεν επιλύεται. Εδώ μιλάμε για 30.000 οικογένειες, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γι' αυτό θα πρέπει να αποτανθούμε στην κυβέρνηση της Ισπανίας. Ωραία. Η κυρία Φαραγκούτ. Πράγματι, η περιφερειακή κυβέρνηση αμφισβητήθηκε και φυσικά και το συνταγματικό ε, δικαστήριο καθώς και τα εθνικά δικαστήρια αποφάθηκαν και είπε ότι αυτό συμβαδίζει με το ρυθμιστικό πλαίσιο, αφορά ε, κρατικές αρμοδιότητες, το θέμα των επιδοτήσεων και ε, είναι αντικείμενο ενός εθνικού διατάγματος ετησίως. Και αυτό αφορά και μία απόφαση, εθνική απόφαση και έτσι έκλεισε η συζήτηση. Άρα εγώ υποστηρίζω την Ένωση αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να πούμε σε ένα κράτος το τι πρέπει να κάνει. Τη στιγμή που τα εθνικά δικαστήρια έκριναν ότι το θέμα έχει καλός, νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Ναι, εδώ μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα. Ναι, μα εγώ βασίζομαι στον εθνικό νόμο. Ναι. <laughs> Μερικές φορές ναι, μερικές όχι. Ροντρίκες, για να διασαφηνίσουμε το ζήτημα. Υπάρχει κρατική αρμοδιότητα και πάντα ανανεώθηκαν οι επιδοτήσεις επιτοκίου. Και ε, όπως μας εξήγησε γραπτός η Ένωση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, παραβίαση των ε, δικαιωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη το ότι πλήττονται δύο βασικές αρχές, η νομική ασφάλεια και η νόμιμη εμπιστοσύνη, γιατί στην ουσία ανανεώνονταν αυτές οι επιδοτήσεις ε, ε, επιτοκίου υπόθηκων δανείων και κάποια στιγμή δεν ανανεώθηκε αυτή η σύμβαση. Άρα, τη στιγμή που κάποιος έμπαινε στη δυναμική αγοράς μιας κατοικίας όπου έρεται ένα πλαίσιο, βρίσκεται σε μια κατάσταση πλήρους ευαλωτότητας, γιατί δεν μπορεί να καταβάλει τους τόκους του δανείου. Και αυτό με στα πλαίσια μεγάλης ανασφάλειας και έλλειψης απασχόλησης. Άρα ε, καλό θα ήταν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφανθεί, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έγινε παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων. Διαφορετικά τώρα η Ένωση θα βρισκόταν ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου και όχι στη δική μας Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά, πράγματι η, Ισπανική κυβέρνηση εξουσιοδότησε την κυβέρνηση της Βαλένθια να ε, προβεί σε αυτή την επιδότηση, η οποία δεν έγινε χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Η Ισπανία θα έπρεπε να το έχει ελέγξει αυτό και δεν το έκανε. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την πτυχή τη στιγμή που μπορώ να παρέμβω κι εγώ θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή Αναφορών να αποστείλει μια επιστολή και στην Κομισιόν και στην Κεντρική Κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό έχετε. Πολύ σύντομα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, παρεμβάσεις ε, όλων των βουλευτών ε, και φαίνεται να στηρίζουν τις αντιπροσωπείες μας που ήρθαν εδώ. Μας εκπλήσει κάπως η παρέμβαση του Ζώπου του Λαϊκού Κόμματος και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί όλες οι αποφάσεις στα ισπανικά δικαστήρια δικαιώνουν τις ενώσεις μας και όχι το κράτος. Η μόνη απόφαση που έχει εκδοθεί είναι αυτή του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία όμως και αυτή είναι υπέρ των ε, δικαιούχων, γιατί ακριβώς άλλαξε το κριτήριο που όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κι εσείς, ε, ε, αποφάσισαν να καταργηθούν όλες οι επιδοτήσεις για κάθε είδος καταλήματος, για κάθε είδος κατοικίας. Γι' αυτό και ακριβώς είμαστε και πήγαμε στους διαμεσολαβητές και σε όλους που είπαν ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το κριτήριο και να σωθούν κάποιοι Με εντυπωσιάζει λοιπόν που το ίδιο το Λαϊκό Κόμμα έχει αναγνωρίσει αυτή τη, εδώ ότι ε, όντως έπρεπε να, κάνει, να γίνει μια νομοθετική αλλαγή ώστε να ανακτηθούν όλα αυτά τα επιδόματα τα οποία καταργήθηκαν σε εκείνη τη φάση. Και από την άλλη πλευρά η Κομισιόν λέει ότι ναι, δεν πρόκειται για οικονομικό μόνο θέμα. Αυτό είναι ένα προϊόν υψηλού κινδύνου. Ε, δεν είναι μάλλον προϊόν υψηλού κινδύνου, είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Εφόσον δεν μπορεί ε, μια χώρα να το τηρήσει, τότε οι πολίτες της Ένωσης, να σας πω, θα χάσουμε την πίστη μας σε αυτό το θεσμό. Μας λέτε ότι δεν είναι δική σας δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε το διάλογο μαζί σας μετά τις ε, απαντήσεις που θα λάβουμε στις επιστολές που θα στείλουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα περνάμε στην επόμενη αναφορά, η αναφορά 273 του 2013 από τη Σλοβακία. Πρόκειται για μια αναφορά σχετικά με τις εργασίες εξόριξης ουρανίου στο Κόσιτσε της Σλοβακίας. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, εκ μέρους των ε, αναφέρατων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δέχεστε σήμερα. Είμαστε κάτοικοι του Κόσιτσε, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στη Σλοβακία. Υπάρχει μια περιοχή για Γιαχόντνα, η οποία είναι πολύ αγαπητή για αναψυχή. Ο κόσμος πηγαίνει, εκδρομές, και περιπάτους. Επίσης υπάρχει και κοίτασμα ουρανίου στην ε, Γιαχότνα, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στου, στις επιγές πόσιμου νερού και στον υδροταμιευτήρα της ε, Γιόχουτνα. Η εξόριξη ουρανίου στο Κόσιτσε έχει πάρα πολλούς κινδύνους και απειλεί και το περιβάλλον αλλά και τους κατοίκους. 113.000 υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί στην αναφορά του 2008 και στο δημοψήφισμα που έγινε οι κάτοικοι της περιοχής ε, αποφάσισαν όχι στην εξόριξη ουρανίου. Παρόλα αυτά όμως το Υπουργείο Οικονομικών της Σλοβακίας και ε, υπέγραψε μια σύμβαση με την Εταιρεία Εκμετάλλευσης των Κοιτασμάτων Ουρανίου για να αρχίσουν εργασίες εξόρυξης. Το 2014 εισήχθη μια τροπολογία στη, στο, νόμο, ε, στο γεωλογικό ε, νόμο που επιτρέπει την εξόρυξη ουρανίου σε ε, προστατευμένες περιοχές, όπως η συγκεκριμένη. Εμείς οι πολίτες θέλουμε να απαγορευτεί πλήρως οποιαδήποτε εξόρυξη ε, με ορυκτών ε, και ουρανίου στην περιοχή, εφόσον θέτει σε κίνδυνο περιβάλλον και ανθρώπου. Οι πολίτες είναι εναντίον της εξόρυξη αυτή. Η κατάσταση βέβαια έχει βελτιωθεί σε σχέση με το 2012 που υπήρξε το απόγειο των εργασιών, όμως δεν ε, σταμάτησε. Εμείς είμαστε εδώ για να σας δείξουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για μας. Αυτό που ε, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση είναι να εξορίσονται ραδιενεργά υλικά στο Κόσιτσε και σε όλη την υπόλοιπη Σλοβακία. Θα ήθελαμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε να υποβάλλετε την αναφορά μας στα άλλα θεσμικά όργανα, τα οποία με τη σειρά τους θα την ε, παρακολουθήσουν και θα την ε, προωθήσουν. Πρέπει να προστατευτεί το περιβάλλον, να προστατευτεί η, νομοθεσία και οι κάτοικοι της περιοχής. Σας κάνουμε έκκληση να πιέσετε το Υπουργείο Οικονομικών να ε, ανακαλέσει αυτό το μνημόνιο συνεννόησης που έχει υπογράψει με την εταιρεία εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων ουρανίου. Οι πρακτικές της εταιρείας αυτής δεν είναι συμβατές με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές του Κόσετσε προσπάθησαν να σταματήσουν τις εξορτικές δραστηριότητες, ωστόσο ε, οι προσπάθειες αυτές έλαβαν τέλος με πρωτοβουλία της κυβέρνησής μας. Θα θεωρούσαμε επομένως ότι ε, στραγγαλίστηκαν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές η βούληση των κατοίκων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Σλοβακίας αυτή τη στιγμή εγκρίνει ε, το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης, διερεύνησης ε, κοιτασμάτων σε άλλες περιοχές της Σλοβακίας χωρίς να ρωτήσει τους κατοίκους. Δεν σέβονται ούτε εμά ούτε το περιβάλλον. Θα σας ζητήσουμε λοιπόν να υποβάλλετε την αναφορά αυτή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στην Αρμόδια Επιτροπή, έτσι ώστε να παρακολουθεί σε την κατάσταση και να διερευνήσει περισσότερα. Και θα θέλουμε επίσης να σας παρακαλέσουμε να καλέσετε εμπειρογνώμονες που θα εκτιμήσουν την κατάσταση και να ε, αναθέσετε μία έκθεση αντικτύπου για τις επιπτώσεις των εξοριστικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και στις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα στον κύριο Μαρτίνα από ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, εκφράσει την άποψη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον αναφέροντα που ε, παρουσίασε νέες πληροφορίες. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι μετά από αυτές τις νέε πληροφορίε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί πως υπάρχει παραβίαση ευρωπαϊκής Νομοθεσία και δεν μας δίνει τη δυνατότητα να ε, θέσουμε σε εφαρμογή κάποιο, ε, κάποια δράση. Υπάρχουν ε, αυτό το θέμα είναι στην αρμοδιότητα των εθνικών αργών, οι οποίες θα αποφασίσουν για το πώς θα διαχειριστούν τα απόβλητα από τις εξορρυκτικές αυτές δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θεωρεί ότι η σωστή εφαρμογή της ε, νομοθεσίας καθιστά δυνατή την κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη εξόριξη ε, ουρανίου. Αυτή είναι η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στα μέλη. Θα ήθελε κάποιος το λόγο. Ζητώ συγγνώμη. Δεν σας γνωρίζω. Είσ... Δεν είστε όμως ευρωβουλευτής, κα... αν δεν κάνω λάθος. Μόνο οι ευρωβουλευτές έχουν το δικαίωμα να συζητήσουν στην αρχή την κάθε αναφορά. Ο κύριος Γιάρη έχει το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να αρχίσω διαφορετικά, να πω ότι καταλαβαίνω απόλυτα το σκεπτικό του αναφέροντος. Υπάρχουν εξωρετικέ δραστηριότητες, υπάρχει κοίτασμα ουρανίου πολύ κοντά στα αποθέματα πόσιμου νερού με κίνδυνο μόλυνσης. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ πάλι γυρίζουμε σε κύκλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δήλωσε ξεκάθαρα. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να φροντίζει να εφαρμόζεται σωστά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όμως εδώ δεν υπάρχει θέμα παραβίασης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και εδώ επανέρχομαι στο ότι είπα γιατί γυρίζουμε σε κύκλους. Εγώ να ρωτιέμαι κάτι άλλο. Πόσο ρεαλιστικό είναι ένα τέτοιο έργο, το οποίο δεν έχει αρχίσει ακόμα. Δεν έχουν αρχίσει εξορρυκτικέ δραστηριότητε. Πόσο ρεαλιστική λοιπόν είναι η έναρξή τους όταν έχει καθυστερήσει τόσο πολύ. Ίσως όταν θα έχει αρχίσει ε, να μπορούμε να το εξετάσουμε καλύτερα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Όμως ε, όταν βρίσκεται ακόμα στο στάδιο του σχεδιασμού εμείς δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε. Δεν έχουν γίνει οι μελέτες που θα μας βοηθήσουν στην αξιολόγησή μας. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Υπάρχει μία σάφια, μία βεβαιότητα η οποία δεν ε, μας βοηθά καθόλου. Ευχαριστώ πολύ. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για να αντιδράσετε σε αυτά που μόλις ακούσατε. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε έχει ως εξή. Η εταιρεία εκμετάλλευσης έχει ολοκληρώσει τη διερεύνηση της περιοχής και τώρα θα υποβάλει την εκτίμηση αντικτύπου και θα κάνει αίτηση για δικαιώματα εξόριξης. Επίσης, θα γίνει και αίτηση για νέες διερευνητικές δραστηριότητες σε μια νέα τοποθεσία. Εδώ πρόκειται για διερεύνηση δυνατότητας εξόρυξης σπάνιων γεών. Και εδώ ε, σε αυτό συμπεριλαμβάνονται ραδιενεργές ε, ραδιενεργά ορυκτά. Έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα ουρανίου. Το μνημόνιο συνεννόηση που έχει υπογραφεί ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Εταιρεία Εκμετάλλευση θεωρούμε πω αποτελεί κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων μας. Εμείς ε, οι πολίτες του Κόσιτς έχουμε απορρίψει, έχουμε καταψηφίσει για την έναρξη των εξορρεκτικών δραστηριοτήτων και ζητούμε από τους ευρωβουλευτές να κάνουν έκκληση στην κυβέρνησή μας έτσι ώστε να ανακαλέσει το μνημόνιο αυτό και να σταματήσει περαιτέρω δραστηριότητε. Οι πολίτε δεν επιθυμούν εξωτικέ δραστηριότητε στην περιοχή. Δεν θέλουμε καν να ξεκινήσουν, διότι εάν ξεκινήσει άλλη αναφορά και περιμένουμε άλλα τρία χρόνια μέχρι να συζητηθεί, πιστεύω πω τότε οι εξωτικέ δραστηριότητε θα έχουν αρχίσει και θα είναι πια αργά. Εάν ζητήσουμε λοιπόν την ε, γνωμοδότηση εμπειρογνωμόνων στην εκτίμηση περιβαλλοντικού αντικτύπου, τότε νομίζω πως θα είναι ο κατάλληλος χώρος και η κατάλληλη στιγμή για την εκτίμησή τους. Δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί η εκτίμηση αντικτύπου τώρα και να τοποθετηθούν οι υπηρεγνώμονες τώρα, όμως πιστεύω πως ε, είναι το πρώτο βήμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να γίνει σεβαστή η επιθυμία των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη Σλοβακία δεν έχει γίνει κάποια κίνηση, δεν έχει υπάρξει κάποια συνέχεια και δεν νομίζω ότι έχει νόημα να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Προτείνω λοιπόν να την κλείσουμε, όμως Πιστεύω πως ε, μπορούμε να στείλουμε μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως μας ζητήσατε και να τους ζητήσουμε να παρακολουθούν τις ε, επόμενες δραστηριότητες της εταιρεία αυτής και επίσης μπορούμε να αποστείλουμε μια επιστολή στη Δημοκρατία της Σλοβακίας όπου θα αναφέρουμε ότι ζητάμε την ε, παρακολούθηση του θέματος και εφόσον διαπιστωθούν κάποιες αλλαγές μπορείτε να κάνετε μία άλλη αναφορά και να τη στείλετε στην Επιτροπή Αναφορών. Το δάχιστες λύση, ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο λοιπόν σημείο που έχουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη είναι η αναφορά 145 του 2012 από τον Χάινο Κριστόφερσον, γερμανικής ηθαγένειας σχετικά με τις αξιορρυκτικές δραστηριότητες στη Λαπωνία και την Ανατολική Φιλανδία. Ενημερώθηκα ότι δεν είναι παρόν ο αναφέροντας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μαρτίνα της Γενικής Διεθνής Περιβάλλοντος, να εκφράσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τοποθετηθεί για την αναφορά αυτή υπήρξαμε πολύ δραστήριοι σε θέματα εφαρμογής ευρωπαϊκού ε, δικαίου, ιδιαίτερα για τις εξορρυκτικές δραστηριότητες στην Φιλανδία. Έχουμε παρακολουθήσει τη ε, διαδικασία μεταφοράς ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τη Φιλανδία και σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάση. Το ίδιο και με τις επίσημε, τα επίσημα αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τις εξορρυκτικές δραστηριότητες στην Ανατολική Φιλανδία. Ζητήσαμε επίσης πληροφορίες για τα ατυχήματα που έχουν συμβεί στο ε, ορυχείο της Ετάβημα. Υπάρχουν προβλήματα νομικά ε, εξαιτίας της κακής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να γίνεται σεβαστή και εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εξορρεκτικές δραστηριότητες δεν θα παραβιάζουν ευρωπαϊκούς νόμους. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Μου φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε τις αναφορές σήμερα. Έχουμε μαζί μας την ε, κυρία Κιλόνεν. Ωστόσο, να σας ενημερώσω, κύριε Κιλόλινεν, ότι ε, δεν έχετε πλήρες καθεστώς θερμηνίας από τα φιλανδικά. Μπορείτε να, ακούσετε, μπορείτε να μιλήσετε φιλανδικά, αλλά όχι να ακούσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο έχει αναφερθεί στο ότι υπήρξαν πάρα πολλέ ε, περιπτώσει παραβίαση Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όχι μόνο στην Ανατολική Φιλανδία, αλλά και στην Τάλιβα, στη Λαπωνία. Μάλιστα, εξορρυκτικέ δραστηριότητες ε, λαμβάνουν χώρα και σε προστατευόμενες περιοχέ του δικτύου Νακτούρα 2000, στο Σάλμινεν, το Κάιλι, το Λούμιερ και το Κίμι Έρβη, ε, αποτέλεσμα της εξορρυκτικής δραστηριότητας είναι η μόλυνση των υδάτων. Τα νερά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πουθενά, ούτε για πλήσιμο ρούχων, ούτε καν στη σάουνα, ούτε για να πλύνεις την αυλή σου. Και προέρχομαι ίδια από την περιοχή αυτή και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι αυτή η εταιρεία έχει δηλώσει επίσημα ότι δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές κάτω από τις οποίες έλαβε την άδεια εξόριξης. Οι περιφερειακές αρχές είναι, ε, που είναι υπεύθυνε και αρμόδιες στο θέμα αυτό δεν αντέδρασαν στο γεγονός αυτό και δεν μπόρεσαν να ζητήσουν ευθύνες από την εταιρεία εκμετάλλευσης. Δηλαδή υπάρχει παραβίαση των υποχρεώσεων των περιφερειακών αρχών. Η μόλυνση των υδάτων και του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής είναι γεγονός το οποίο συνιστά περιβαλλοντική καταστροφή και ε, έχει και άλλες επιπτώσεις. Απειλείται όχι μόνο το περιβάλλον, όχι μόνο οι περιοχές του δικτύου Natura 2000, αλλά και η τοπική κουλτούρα των ε, Σάμι, του, του αυτόχθονου πληθυσμού εκεί και της ε, εκτροφής ταράνδων στην οποία δραστηριοποιούνται. Υπάρχει παραβίαση του άρθρου 38 στην συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχει γίνει μελέτη αντικτύπου των εξορρυκτικών δραστηριοτήτων ε, και στην κουλτούρα και την ε, γλώσσα του ε, Σάμι. Δεν έχει γίνει καμία μελέτη για το αν θα είναι στο μέλλον σε θέση να ψαρεύουν, να εκτρέφουν τα ζώα τους και να συνεχίσουν να ζουν την ζωή τους με το παραδοσιακό τρόπο που ζουν μέχρι σήμερα. Μάλιστα, έχουν γίνει προσπάθειες αποδυνάμωσης της νομοθεσίας. Έχουν γίνει προσπάθειες αποχαρακτηρισμού ορισμένων ε, περιοχών από προστατευόμενες σε μη προστατευόμενες. Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι, τοπικές αρχές είναι οι συνυπεύθυνες για το τι συμβαίνει. Δεν έχει αναλυφθεί καμία ευθύνη για προστασία του περιβάλλοντος σε αυτήν την περιοχή. Η περιοχή που όχι μόνο είναι προστατευόμενη, αλλά και ε, ανήκει στους ε, Σάμι. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και με κάνει να ανησυχώ ιδιαίτερα οι παραβιάσεις ε, γίνονται ενάντια στο περιβάλλον και ενάντια στην ε, νομοθεσία, στα δικαιώματα των πολιτών, στα θεμελιώδη δικαιώματα. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι η Τάλβη Βάρα είναι μόνο ένα παράδειγμα άδεια που έχει δοθεί για να διοχετεύονται απόβλητα στο νηδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Τα απόβλητα από την επεξεργασία ουρανίου καταλήγουν λοιπόν σε νερό που πηγαίνει στο περιβάλλον. Εάν δεν ασχοληθούμε με αυτό το θέμα που απειλεί τη φυσική ισορροπία, απειλεί την υγεία των ανθρώπων, τότε ε, θα ε, έχουμε τρομακτικές επιπτώσεις. Τώρα, σχετικά με την προστασία των υδάτων, πρέπει και εδώ να δείξουμε μεγάλη προσοχή και να είμαστε επάγρυπνοι. Το, τα ύδατα αποτελούν και πηγή απασχόλησης για πάρα πολλούς πολίτες, ξέρετε, και η ζημιά που γίνεται είναι ανεπανόρθωτη. Ο κύριος Γιάρη έχει το λόγο. Ο πρόεδρος ε, νομίζω είπε αυτό που θεωρώ και εγώ πως μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά. Θα ευχαριστήσω λοιπόν την συνάδελφη από τη Φιλανδία που τοποθετήθηκε και θα προτείνω να καταγραφούν στα πρακτικά όλα αυτά που είπατε και προτείνω σε αυτή την περίπτωση να αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή και να ζητήσουμε μια επίσημη απάντηση. Είχα αρχικά την εντύπωση ότι μπορούσαμε να την κλείσουμε όπως και εσείς, αλλά μετά από αυτά που άκουσα νομίζω πως καλύτερα να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή, να καταγραφούν αυτές οι λεπτομέρειες στα πρακτικά και να ζητήσουμε ε, εξηγήσει, ίσως όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά από τις φιλανδικές αρχές. Αυτό λοιπόν θα έλεγα, να αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή και να αναμένουμε νεότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ. Yes, So thank you very much. I, accept your position, Peter. Um, we keep open this. Μάλιστα, συμφωνώ, Πίτερ. Θα κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή. Θα ζητήσουμε απάντηση από τις ε, φιλανδικές αρχές σχετικά με αυτά που μας είπατε και θα σας κρατήσουμε ενήμερους για την πρόοδο της κατάστασης σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν κάνω λάθος, τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλό σας βράδυ και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Καλό βράδυ.